Mes chers collègues, euh, Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα να μας συγχωρείτε που καθυστερήσαμε την έναρξη της συνεδρίασης. Αλλά έπρεπε να έχουμε κάποιες ε, αλλαγές στο πρόγραμμα. Να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Οπότε χρειάστηκε να συντομεύσουμε τη διάρκεια της συνεδρίασης. χθε ούτω ή άλλω ενημερωθήκαμε, οπότε γι' αυτό σα ειδοποίησαμε και εσά καθυστερημένα. Για το πρώτο σημείο, έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Έχετε δει το σχέδιο ημερήσια διάταξη στο δελτίο τη Επιτροπή μα. Έχω κάποιε διευκρινήσει απλώ να σα επισημάνω για την ψηφοφορία για τις εκτιμήσεις, το προσχέδιο για την κατάσταση προβλέψεων των, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία αυτή αναβάλλεται, διότι το Προεδρείο δεν έχει ακόμα εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων. Ο εισηγητής είναι στη διάθεση της ε, Επιτροπής Προβλεσμών για να ενημερώσει για το πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις το απόγευμα και οι συντονιστές θα το συζητήσουν μετά την συνεδρίασή μας μετά το πρωί. Κατά τα άλλα, σκεφτήκαμε να συμπεριλάβουμε στην ημερήσια διάταξη μια μελέτη σχετικά με τον τρόπο που τα κράτη-μέλη συντονίζουν και χρησιμοποιούν τι συνεισφορές προ τον ευρωπαϊκό ε, προπολογισμό με τους εθνικούς προπολογισμού. Μετά από αίτηση των ε, δύο ε, εισηγητών, της κυρίας Γένσον και του κυρίου Τονκάν, δεν θα γίνει η παρουσίαση, διότι τα έγγραφα που ετοιμάστηκαν δεν ήταν ικανοποιητικά και δεν ικανοποιούσαν την αρχική πρόθεση να ενημερωθούμε. Τώρα, τέλος, οι δύο εισηγητές για τα δημοσιονομικά έτη 2004, η κυρία Γένσεν και για το 2015, η κυρία Χάιντερ. Και θα περιμένουν να δούμε πρώτα να κάνουμε πρώτα την ακρόαση με τους δύο επιτρόπους για την κατάσταση των αναγκών πληρωμών στην Ένωση, την γενική κατάσταση και ιδίως ό,τι αφορά την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια εκδοτική βοήθεια 11 δις ευρώ προς την Ουκρανία και η κατανομή της βοήθειας αυτής έχει προκαλέσει πολλές απορίες. Έχετε όλοι λάβει το σχέδιο προφορικών ερωτήσεων μοιράστηκε χθε σε όλου. και σήμερα το απόγευμα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για το περιεχόμενο τη προφορική ερώτηση. Άλλη αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Γένσεν, που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα το πρωί, ζήτησε το σημείο που την αφορά για το σχέδιο διευθυντικού προπολογισμού, αριθμός 1, στον Γενικό Προπολογισμό του 2014, να το δούμε το απόγευμα. Και Αντιστρόφως, η κυρία Γκρέσλε, που είναι στην πρώτη σειρά πάντοτε χαμογελαστή, δυναμική και αποτελεσματική, ζήτησε το σημείο 17 και 18 του προβλέπονταν για σήμερα το απόγευμα να τα συζητήσουμε σήμερα το πρωί. Αυτά. Η Αίντερ Γκαντιασάμπαλ θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι ο Πρόεδρος Πάντα συνήθως λέει χρόνια πολλά για διάφορα γενέθλια και έκτακτες περιστάσεις. Και θα ήθελα ε, να του ευχηθώ να του ζήσει το παιδί του γιατί έγινε πατέρας ε, πρόσφατα και σήμερα είναι και η μέρα του πατέρα στην Ισπανία, 19 Μαρτίου. Ε, συγχαρητήρια. Ε, να σας ζήσει και ελπίζω το βράδυ να σας αφήνω να κοιμάστε τα μπιμπερό και τα διάφορα ξυπνήματα και κλάματα του μωρού και να μπορείτε και να ξεκουράζεστε λίγο, να σας ζήσει το παιδάκι σας. Ευχαριστούμε, Ειντερ. Είναι πολύ συγκινητικές οι ευχές σου αυτές, προσωπικές ευχές. Είμαι σε ηλικία να είμαι και παππούς βέβαια, κάτι που ούτως ή συμβαίνει, με επτά εγγόνια ο, των ο ένας είναι 8 ημερών. Είναι προφανώς μια, ένα ευτυχές γεγονός για τη ζωή του ανθρώπου και ο καθένας μας στην οικογενειακή του ζωή έχει ευτυχώ τέτοιε ευτυχισμένε στιγμές που είναι και πιο σημαντικέ από την πολιτική μα δράση. Να επιστρέψουμε όμω στα πολιτικά ε, πράγματα. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Έντερ. Ε, και τους ευχόμαστε όλοι να ζήσει τέτοιες ευτυχισμένες στιγμές. Την θαυμάζω. Και είχα την ευκαιρία ως πατέρας να παραστώ στον, στην εγκυμοσύνη και την, τον ροκετό της ε, γυναίκας μου, οπότε ξέρω πώς τη συναισθήματα μπορεί να έχει μια γυναίκα που πρόκειται να γίνει μητέρα. Αυτά για το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Για τις ανακοινώσεις του Προέδρου τώρα. Θα το είδατε στο δελτίο της Επιτροπής μας, στο ενημερωτικό δελτίο, να σας ανακοινώσω μια σημαντική ημερομηνία. Θα ξέρετε ότι για την ενδιάμεση περίοδο, για το τέλος δηλαδή της θητείας, για το διάστημα μεταξύ των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου και την ανάλυση καθηγόντων από το νέο κοινοβούλιο την 1η Ιουλίου, προβλέψαμε μια έκτακτη συνεδρίαση τη Επιτροπή Προπολογισμών για να ακούσουμε τον Επίτροπο που ασχολείται με τους προπολογισμού εσύ βάσει των υιοθότων τον προπολογισμό για το 2015 που μπορεί να εγκρίνει το Σωμά των Επιτρόπων. πριν την ε, επίσημη παρουσίασή του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ε, κοινή γνώμη. Αρχικώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι αυτό θα γινόταν στις 4 Ιουνίου, τελικά όμως αναβλήθηκε για μια εβδομάδα. Οπότε να το σημειώσετε παρακαλώ, αλλά θα σας το επιβεβαιώσουμε γραπτός. 11 Ιουνίου, Τετάρτη 11 Ιουνίου, το Σώμα των Επιτρόπων θα εγκρίνει το σχέδιο προπολογισμού για το 2015, οπότε το δεύτερο μισό του πρωινού εκείνη της ημέρας θα έχουμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση για να ακούσουμε τον Επίτροπο. Με την ευκαιρία αυτή να σας ε, επαναλάβω και να σας θυμίσω ότι αφού θα είναι η τελευταία μας συνεδρίαση να γιορτάσουμε μαζί τα πέντε χρόνια δουλειάς που έχουμε κάνει μαζί και να αποτίσουμε φοροτιμής σε όλες και όλους που συμμετείχαν Ίσως να χρειαστεί να θυμηθούμε και κάποιες δύσκολες στιγμές ή κάποιες δραματικές στιγμές που έζησαν κάποιοι ε, συνάδελφοι στις οικογένειές τους και με τους ε, συνεργάτες μας εδώ και με άλλους ε, εργαζόμενους θεσμικά όργανα. Νομίζω λοιπόν ότι στις 11 Ιουνίου θα είναι μια καλή ευκαιρία για να γιορτάσουμε, να πιούμε και λίγη σαμπάνια και να συγχαρούμε όσους έχουν επανεκλεγεί ή να αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους που θα μας αφήσουν. Για τις υπόλοιπες τώρα ανακοινώσει. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 4ης Μαρτίου. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις ως το τέλος της συνεδρίασης, θεωρούμε ότι τα πρακτικά αυτά είναι εγκεκριμένα. Τώρα, εάν είναι εδώ ο ενδιαφερόμενος και είναι ο συνάδελφος Νταρντέν, να ξεκινήσουμε με τα σημεία 7 και 8. Συνάδελφο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σχετικά σύντομος. Θα σας παρουσιάσω αυτά, αυτές τις δύο κινητοποιήσεις που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και τελευταίες της θητείας μας. Μία λοιπόν ε, στα πλαίσια μιας εταιρείας ε, μεγάλων επενδύσεων στην Ιταλία που ζητάει 3 εκατομμύρια για 1.140 ε, απολυμμένους, πάνω από 3 εκατομμύρια μάλλον για 1.140 σε βάση το άρθρο 2 του προηγούμενου κανονισμού, γιατί ακόμη βασιζόμαστε για το προηγούμενο κανονισμό για την, με το κριτήριο της παγκοσμιοποίησης ε, και έχουμε φτάσει σε όριο τέσσερων μηνών τους 500 ε, απολυμμένους. Θέλετε να συνεχίσω, Πρόεδρε, και με το επόμενο. Η δεύτερη κινητοποίηση σχετίζεται με αίτημα για 1.965.000 για 285 απολυμμένες από 15 εταιρείε ε, ε, στην Ανδαλουσία και πρόκειται και πάλι για το κριτήριο της κινητοποίησης ε, και πάλι εγγράφεται στα πλαίσια του προηγούμενου κανονισμού. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Έχουμε καλέσει το την κυρία Μωγάν Σαθία που είναι η συγγήτρια από την Επιτροπή Απασχόλησης για να μετάσχει στις συζητήσεις μας, αλλά δεν έχει καταφτάσει από ό,τι βλέπω. Και θα μετάσχει και στην ομάδα παρακολούθησης Monitoring Group ε, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Ε, σε σχέση με αυτά που μας είπε ο εισηγητής μας, έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις? Όχι, ωραία. Όπως το είπε, υπαγόμαστε στο καθεστώς του προηγούμενου κανονισμού και ως προς το χρονοδιάγραμμα η καταληκτική για τι τροπολογίε είναι στι 12 το μεσημέρι 24 Μαρτίου, στην Επιτροπή Απασχόληση ψηφοφορία στι 18 Μαρτίου και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών 1η Απριλίου. Με στόχο, έγκριση από την Ολομέλεια προτού εκπνεύσει η απριλιου με στοχο εγκριση απο την ολομελεια πρωτου εκπνευσει η θητεια ε, στο Στρασβούργο. Αυτό ισχύει και για τα δύο θέματα. για το Ιταλικό και για το Ισπανικό πρόγραμμα. Ε, θα πρότεινα τώρα στην Ίγκε να μας παρουσιάσει τα θέματα 17 και 18. Ίγκε. Ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσω από τα πολιτικά κόμματα. Να σας πω πώς έχουν οι διαπραγματεύσεις. 4 Μαρτίου συναντήθηκαν οι σκιώδεις ηγητές και συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει γρήγορα ότι θέλουμε να συμφωνήσουμε το Συμβούλιο. Είμαστε τμήμα της λύσης και όχι τμήμα του προβλήματος. Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων την περασμένη Τετάρτη ε, ματαιώθηκε γιατί ματαιώθηκαν οι πτήσεις από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο. Προσπάθησα ε, εν ώψη ε, της επόμενης συνεδρίασης που είναι αύριο το πρωί με email να επιτύχω μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει γενική συνένεση για το κείμενο. Το κείμενο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ΑΦΚΟ. Ε, ε, το θέμα του ελέγχου των λογαριασμών εκκρεμεί ακόμα, αλλά βρήκαμε ε, μια λύση και εκεί για εξωτερικούς ελεγκτές. Το έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο διακομματικά. Μέχρι τώρα το Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί επί του κειμένου που έχουμε εκπονήσει εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και χτες το βράδυ δυστυχώ μα διαβίβεσε ότι δεν έχει και εντολή. Οπότε αύριο δεν θα θεωρηθεί τριμερή διάλογο η συνάντηση, απλή ανταλλαγή απόψεων θα είναι. Πάντω εγώ πιστεύω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και μπορούμε άτυπα να συμφωνήσουμε τα τρία όργανα και στι 25 Μαρτίου μπορεί η Κορεπέρ να το επιβεβαιώσει αυτό. Τουλάχιστον αυτή είναι η επιθυμία μας και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μπορέσει αυτό αύριο να συμφωνηθεί. Είναι σε καλό δρόμο. Πράγμα που δεν μπορώ να πω για το δεύτερο θέμα φυσικά. Να συνεχίσω έτσι με το επόμενο. Να σταματήσω εδώ, Πρόεδρε, να συνεχίσω για να σας πω και για το 18. Το δεύτερο λοιπόν είναι ε, η διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, Connecting Europe. Ε, είναι δύσκολο αυτό το θέμα εδώ γιατί το Συμβούλιο τα έχει στυλώσει για να το πω έτσι και συνεχίζει να μπλοκάρει τα πράγματα. Χτες ε, είχα μια συνομιλία με τον Έλληνα πρέσβη προεδρεύοντα και το Γενικό Διευθυντή Ζωζό για να τους ε, βολιδοσκοπήσω λίγο προς τα που το πηγαίνουν. Για πόσα χρόνια καλύπτονται οι μεταφορές πιστώσεων και πώς θα γίνονται, με ποια διαδικασία και με ποιους όρους και προϋποθέσεις. Σε αυτό το σημείο παραμένουν τα πάντα ακόμα ανοιχτά. Θα ήθελα να μας δώσω μια συμβολή, να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, αλλά πρέπει να κινηθεί εκείνο πρώτα. Στο άρθρο 178 έχουμε προβλέψει επιπλέον βελιξία ε, ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε περίπτωση που δεν περάσει θα ήταν πολύ λυπηρό αυτό επί της ουσίας. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα πρέπει να σας πω ε, Κανονικά το Συμβούλιο πρέπει να μετακινηθεί. Και αν δεν αλλάξει στάση θα πάνε χαμένα πολλά χρήματα από το Connecting Europe. Και δεν μας ε, συμφέρει ούτε εμάς αυτό. Θέλουμε εξυγχρονισμό. Ε, στην Ευρώπη και αυτά που λέγουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι κενό γράμμα και δεν ισχύουν για τις διοικήσεις. Διατρανώνουν διάφορα μεγαλόστομα και τώρα τα Υπουργεία Οικονομικών, ορισμένα τμήματα και υπηρεσίες μπλοκάρουν αυτά. Και μάλιστα με ιδιαίτερη χαρά. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συμφωνήσουμε. Καλό θα ήταν να καταλάβει και το Συμβούλιο ότι είναι λεφτά για τις χώρες. Θέλουμε μια πιο σύγχρονη Ευρώπη. Και τελικά τα κράτη-μέλη τι κάνουν. Τρεκλοποδιά στον εαυτό τους βάζουν. Δεν τα έχω καταλάβει όλα σε αυτή την υπόθεση, αλλά μπορεί και να μην χρειάζεται κιόλα να μην είναι δική μου δουλειά, να τα καταλαβαίνω. Έτσι έχουν τα πράγματα και πάλι σήμερα το βράδυ θα τα συζητήσουμε και ελπίζω να βρούμε ένα δρόμο, να προχωρήσουμε. Αύριο θα ξανασυνεδριάσουμε και ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, σύντομα να δοθεί το πράσινο φως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ίγκε. Ξεκάθαρο όλα αυτά που μας είπες, κρίκια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα με την ιδιότητα του εισηγητή για τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη να αποφανθώ κι εγώ διότι έλαβα γνώση κι εγώ των δυσκολιών συγγνώμη, που <laughs> ανέφερε Ίγκε. Ε, λοιπόν, για τον δημοσιονομικό κανονισμό, για αυτή τη χρηματοδοτική διευκόλυνση, οι αλλαγέ που προτείνονται αλλοιώνουν σε μεγάλο βαθμό τον κανονισμό όπω εγκρίθηκε. Δηλαδή, πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και σα υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο από πλευρά αριθμών είχε υποχωρήσει από 50 δι, έφτασε τα 33 παρότι ήταν πιεστικό το Κοινοβούλιο στο αίτημά του για αυξημένες επιστώσεις, ε, ούτως ώστε να μπορέσει να δράσει μέσα του προϋπολογισμού για να τονώσει την ανάπτυξη. Είναι στρατηγική σημασία δηλαδή το ζήτημα. Θα ήθελα μόνο να τονίσω πως οι θέσεις του Συμβουλίου από πλευράς ε, δημοσιονομικού κανονισμού είναι τέτοια φύση ώστε να αλλοιώνεται σοβαρά η φύση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Δεν πρόκειται για τεχνικά ζητήματα δημοσιονομικού κανονισμού. Δεν πρόκειται ε, για επίλυση κάποιων αφιλεγόμενων ε, σημείων ε, σε συνεργασία με τους Υπουργούς Οικονομικών. Ε, πάνω κάτω περικόφτουμε περαιτέρω τη χρηματοδοτική διευκόλυνση και δεν επιτρέπουμε ευέλικτη χρήση αυτού για τους φορείς εκμετάλλευσης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα, διότι, ξαναλέω, είναι διαρθρωτικό σημείο, δομικό σημείο αν θέλετε, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και η διευκόλυνση συνέοντα ε, την Ευρώπη, αν δεν αλλάξει η θέση του Συμβουλίου, θα βρεθεί ε, σε μια θέση όπου θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει χρήση του από τους φορείς εκμετάλλευση των προγραμμάτων. Ε, Δεδομένες της φύσης των προγραμμάτων χρειάζονται μακρύτατες προθεσμίες, ώστε να γίνει επιχειρησιακό ένα πρόγραμμα και ως εκ τούτου, αν η θέση του Συμβουλίου περικόψει περαιτέρω τις προθεσμίες και χαθούν τα κονδύλια, τι σημαίνει αυτό περικόπτουν την περαιτέρω κονδύλια στον προπολογισμό και άρα ε, καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση του προγράμματο. Αυτό καταδεικνύει πω η θέση του Συμβουλίου είναι να επανέλθει ε, με διάφορου τρόπου, ε, να αναθεωρήσει μάλλον με διάφορου τρόπου τα συμπεφωνημένα ποσά του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου μέσω παραδείγματο χάρη τη ενημέρωση ή διορθωτικών δράσεων στον προπολογισμό και ούτω ή δεν μα είχε ικανοποιήσει ο προπολογισμό όπω είχε εγκριθεί, αλλά τώρα πια είναι απαράδεκτο. Βλέπουμε με ποιο τρόπο ο δημοσιονομικό κανονισμό ε, ε, αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευση, μεθόδευση και χειραγώγηση από πλευρά του Συμβουλίου. Ε, Ε, ε, ε, το έχουμε ήδη, έχουμε ήδη υπερασπιστεί τη θέση σε διάφορες, από πλευρά διάφορων επιτροπών ενώπιον το Συμβουλίου, αλλά πραγματικά θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα και πόσο κακές είναι οι εξελίξεις που ε, ε, θα επισύρει μια τέτοια αλλαγή αυτή που επιδιώκει το Συμβούλιο. Δεν ε, είναι σωστό να λειτουργεί έτσι το Συμβούλιο και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουμε τελικά να μην καταλήξουμε συμφωνία προτού λήξει η θητεία. Αυτό, ο κίνδυνος ελοχεύει. Ρικέ. Ε, μα ε, το Συμβούλιο το χρησιμοποιεί αυτό ακριβώς ε, για να επιτύχει τους στόχους του. Ο Πρόεδρος, ναι, σε αυτό έγκυται και το πρόβλημα, καταλαβαίνω πολύ καλά. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις. Ε, όχι, ευχαριστούμε την Ίγκε. Τουλάχιστον είμαστε τυχεροί που είναι η συγγήτρια γκε, γιατί είναι τόσο σημαντικό και τόσο λεπτό αυτό το ζήτημα διότι τη χαρακτηρίζει αυτή, αυτός ο δυναμισμός και αυτή η ενέργεια που όλοι γνωρίζουμε. Σα προτείνω να περάσουμε στο σημείο 10, ομάδα παρακολούθησης για την ε, βοήθεια μέσα του Ταμείου για τους Απόρους. Ε, και την εφαρμογή των επιπλέον ε, ποσών που, για το 2014 που έγινε ή θα γίνει. Ε, ξέρετε ποια αρχή διέπει τη λειτουργία των ε, ομάδων παρακολούθησης. Είναι ευκαιρία για μας, ε, για τους εισηγητές και άλλα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού να κάνουν ανταλλαγή απόψεων με αυτούς που έχουν αναλάβει τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου ανακοίνωσαν πως η γάμα δέτα απασχόληση σε γεωργίας ε, ενέργειας ε, η κυρία Γεωργιάνα του Σίσκοβα που είστε εδώ καλωσορίσατε ε, Μανουέλ Γκίφνερ, Έρχονται οι δύο κυρίες. Ο κύριος Σέρς Λεγκάλ ε, για τον ε, διοργανικό συντονισμό. Είστε και εσείς εδώ. Και ο κύριος Πατρίκ Μαλεζά που είναι και επικεφαλής της ομάδας του κλιμακίου. Ε, TG Agri, Arpad Σαμπόλτς, δεν παραφθείρο, τέλο πάντων δεν ξέρω, market officer είστε εσείς. Ε, προϋπολογισμούν ε, Καταρζίνα Ρούσκα, υπάλληλο του τμήματος προϋπολογισμών, εδώ είστε, μας χαμογελάτε, πολύ ωραία. Και η κυρία Λετήσια Γκέρλι, βοηθός. Λετήσια, καλώς ήρθατε. Αυτή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε προσκαλέσει ε, μέλη από την Επιτροπή Απασχόλησης του Κοινοβουλίου και ε, θα έρθει η κυρία Μωγάν Σαχτιέ και θα έρθει εδώ ως αντιπρόεδρος που είναι, εδώ δίπλα μου. Έχουμε δύο εισηγητέ για τον προπολογισμό 2014 και για το 2015. Θα έρθει και η Αν Γένσεν, η Έιντερ είναι εδώ ήδη. Έιντερ, ε, θέλεις να ξεκινήσεις εσύ τη συζήτηση, την παρουσίαση. Ναι. Βεβαίω προφανώς αυτό που έχει σημασία να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να του κάνουμε και ερωτήσει. Θα ήθελα απλώ να εξηγήσω γιατί αποφασίσαμε να ε, συστήσουμε αυτή την ομάδα παρακολούθησης, monitoring group ονομάζεται. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το είδος ε, βοήθεια στο Ταμείο για τη βοήθεια προς τους απόρους. Το έχουμε παρακολουθήσει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας και ήταν ένα από τα προγράμματα ε, που έγινε και συζήτηση και διακύβευμα στο πλαίσιο και της προοπτικές γιατί ήθελαν τα κράτη-μέλη να μειώσουν τη χρηματοδότηση και εμείς αν μη τι άλλο θέλαμε να διατηρήσουμε το ίδιο ποσό και να λειτουργήσει καλά το Ταμείο διότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή που είναι περισσότερο απαραίτητο από ποτέ έπρεπε να ξέρουμε πώς λειτουργεί. Γι' αυτό φτιάξαμε αυτή την ομάδα εργασίας, πώς γίνεται στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο με τους νέους κανόνες, με συμμετοχή ε, ενός ε, τμήματος ε, του Ταμείου Συνοχής, το 1 δις δηλαδή, που αντλούν από εκεί, πώς το διαχειρίζονται, πώς λειτουργεί, υπάρχουν καθυστερήσεις, ολιγορίες. Είναι γεγονός ότι επειδή άργησαν οι διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές και το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο, υπήρξε καθυστέρηση, αλλά το Κοινοβούλιο επέμεινε πάρα πολύ να υπάρξουν μεταβατικά μέτρα για να μην ε, μείνει ε, χωρίς ε, χρηματοδότηση, ο κόσμος που εργάζεται, οι διάφορες τράπεζες τροφίμων και τα Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, δεν έπρεπε να υπάρξει κενό στη χρηματοδότηση ε, λόγω της μεταβατικής περίοδου. Αυτό που θέλω να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια είναι τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει, ποια είναι οι πιθανές λύσεις και πώς βαίνει η λειτουργία αυτού του ταμείου. Ε, Ευχαριστούμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιος θέλει το λόγο. Κυρία μου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Επίτροπος καλωσορίζει την θέση σε ισχύ του κανονισμού στις 11 Μαρτίου για το Ταμείο Βοήθειας προς τους ε, πλέον απόρους και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τη στήριξη του προς αυτό το σημαντικό εργαλείο για να εκφράσουμε την Ευρωπαϊκή Ελληνική με την πρόσφατη έγκριση του κανονισμού. Ο στόχος είναι τώρα να πετύχουμε τη γοργή υλοποίηση και θέση σε του Ταμείου και καταλαβαίνουμε από τι ερωτήσει που λάβαμε από τα μέλη τη Επιτροπή σα, ότι αυτό θεωρείτε και εσεί τη βασικότερη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Έχετε λάβει και κάποιε γραπτέ απαντήσεις, αλλά θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ε, τονίσω κάποια από τα βασικά σημεία. Πρώτα απ' όλα για τον προγραμματισμό. Τα κράτη-μέλη βάσει του κανονισμού έχουν ένα εξάμεινο για να υποβάλουν τα επιχειρησιακά του προγράμματα και να περάσουν στη φάση συνομιλιών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι νομική απέτηση. Ελπίζουμε όμως ότι τα κράτη-μέλη ήδη εργάζονται και ότι αυτοί που έχουν χρησιμοποιήσει το τρέχον εργαλείο για την ε, βοήθεια στα τρόφιμα βάσει και των ε, κονδυλίων της Γεωργίας θα προχωρήσουν γοργά και θα λάβουμε γρήγορα τα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Ήδη είμαστε σε επαφή με κάποια κράτη-μέλη που έχουν προχωρήσει πολύ και ελπίζουμε ότι τα επιχειρησιακά του προγράμματα θα αποβληθούν μέσα στι προσεχεί ημέρε, τουλάχιστον στο τέλο Μαρτίου. Για την ώρα δεν έχουμε λάβει πάντω επισήμω κανένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τα κράτη-μέλη, ωστόσο, δεν χρειάζεται να περιμένουν την επίσημη υποβολή ή έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για να ξεκινήσουν να εφαρμόζουν τόσα προβλέπει το Ταμείο. Χάρη και στην στήριξη του Κοινοβουλίου, ο κανονισμό προβλέπει έναρξη ισχύω την 1η Δεκεμβρίου του 2014 για την ρεσιμότητα για τις δαπάνες, για την επιλεξιμότητα για τι δαπάνες. Και έχουμε λάβει ενδείξει από τα κράτη-μέλη ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες των ε, δημοσιοπρομηθειών για να προβλεφθούν τα απαραίτητα τρόφιμα που περιλαμβάνονται στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Σε συνδυασμό με την παράταση της περίοδου εφαρμογής 2013 και του ετήσιου προγράμματος διανομής τροφίμων για τους πλέον απόρους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εδώ έχουμε τις προποθέσει για να αποφύγουμε τις ε, διακοπές διανομής τροφίμων προς τους πλέον απόρους. Τα κάτι μέλη που έχουν ήδη κάποια πείρα με την επισητιστική βοήθεια είναι αρκετοί αυτοί που ήδη χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό, θα προχωρήσουν πιο γρήγορα. Κάποιοι έχουν προτιμήσει όμω το πρόγραμμα τη ε, κοινωνική συμμετοχή, όπω ονομάζεται, το επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινωνική συμμετοχή, το ΟΠΙΤΟΥ. Ε, οπότε θα προχωρήσουν διαφορετικά. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη και ελπίζω ότι τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα θα υποβληθούν εντό τη διορία του εξαμήνου, δηλαδή 11 Σεπτεμβρίου. Και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα να εγκριθούν με απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω το τέλο τη χρονιά. Ω προ τη διαδικασία έγκριση τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε εφόσον τα διαθέσιμα κονδύλια δεν αρκούν για να καλυφθεί η προχρηματοδότηση του 11%. Οι τιμήσεις για τον προπολογισμό βασίστηκαν στις χαμηλότερες ε, προβλέψεις για τον απαραίτητο προπολογισμό, 2,5 δις ευρώ, ενώ τώρα έχουμε φτάσει στα 3,4 δις για, συνολικό για το συνολικό κόστος. Στο παράρτημα 3 του κανονισμού έχουμε συμπεριλάβει τα κονδύλια με κράτος μέλος και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένα πρόσθετο δις ευρώ από, ευρωπαϊκά, από ευρωπαϊκούς πόρους. Για το ΦΕΔ ήδη έχει γίνει η απαραίτητη. Για το έχει γίνει ήδη μια απαραίτητη πρόσληψη και ευχαριστούμε που ενέκρινε και το Κοινοβούλιο την του προγραμματισμό για αυτό το εργαλείο. Να ολοκληρώσω λέγοντα ότι πέραν από την σύντομη υλοποίηση και τον προγραμματισμό αυτό, το, η Επιτροπή παρακολουθεί και τη διάσταση τη παρακολούθηση. Προκειμένου λοιπόν να έχουμε σωστή συλλογή δεδομένων ευθύ εξ αρχή, γιατί είναι σημαντικό για μα να ξέρουμε ακριβώ πόσα θα δαπανηθούν και πόσοι ακριβώ άνθρωποι θα στηριχθούν, έχουμε ήδη ειδοποιήσει το Κοινοβούλιο και έχουμε κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο την έγκριση στι 13 Μαρτίου κατά εξουσιοδότηση πράξη, η οποία περιλαμβάνει διατάξει για τα δεδομένα που θα πρέπει να συλλέγονται και θα κρατώνται, θα, σε, θα, τηρούνται, θα τηρούνται σε αρχαίο τα κρατημέλη και για την υποβολή εκθέσεων προς το ε, Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία μου. Άλλη παρέμβαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, ε, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας είναι εδώ. Ίσως θέλετε κι εσείς να πείτε κάτι. Να μας πείτε τη δική σας άποψη. όχι. Ωραία. Από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών ούτε. Ούτε εσείς. Κύριε Πρέζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια ευκαιρία αυτή ώστε οι υπηρεσίες μας να εξηγήσουν το πώς θα γίνει η υλοποίηση του πράγματος αυτού. Η δική μας Γενική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την σωστή κατανομή, αλλά για το 2014 έχει ολοκληρωθεί η δική μας δουλειά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Στο μεταξύ, η κυρία Μωράν Σαρτιέ, η συγγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης, κατέφτασε. Σας καλωσορίζω, καλημέρα σας. Θα ήθελες να κάνεις τη δική σου παρέμβαση και να πεις τη δική σου άποψη. Γιατί πέραν από την Έιντερ Κακτία Σαμπάλ που είναι η συγκεκριά μας για το βασικό προπολογισμό το 2015 έχουμε εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμών, Γεωργίας και Απασχόλησης. Και την κυρία Γένσεν, ε, για, το, για τον προπολογισμό μας του 2014 που πρόκειται να έρθει που να είναι. Ελίζαμπετ, Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητέ Έλα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Προπολογισμών. Διότι το να προασπιστούμε το Ταμείο ε, Βοήθειας προς τους πλέον απόρους και από πολιτική σκοπιάς δεν ήταν κάτι το δεδομένο. Επειδή ακριβώς οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είχαν την δική τους άποψη για τα πράγματα. Ξέρω πόσο η Επιτροπή Προπολογισμών και εσύ ο ίδιος Αλέν, εάν μου το επιτρέπεις, αγαπητέ μου πρόεδρε, με τη δράση σου και με τη δική σας δράση ήσασταν ιδιαίτερα αποτελεσματική για την προάσπιση του Ταμείου αυτού. Τώρα, να απευθυνθώ στους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που και εκείνη μας βοήθησε πολύ ε, προς αυτό το στόχο. Ο Έλμερ Κοστέλο, ε. η Έλμερ Κοστέλο ήταν η συγγήτρια για το ΦΕΑΝΤ Έχω συνεργαστεί στενά μαζί τη, γιατί εγώ ήμουν υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οπότε ήταν σαφή ε, ήταν σαφής ο αλληλοσυγχυντισμός των δύο. Δύο λόγια μόνον. Να πω ότι από πολιτικής σκοπιάς το όλο αυτό θέμα ήταν πολύ σημαντικό και ζωτική η βοήθεια της Επιτροπής Προπολογισμών, κυρίως μετά από όλες τις ενέργειές μας, προκειμένου να εκφραστεί οικονομικός η αλληλεγγύη μας ε, εξαιτία της κρίσης. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών είναι κάτι που προσδοκάται πραγματικά διακαώς, διότι η ευρωπαϊκή βοήθεια προς τους πλέον απόρους είναι απολύτως αναγκαία. Σήμερα πάνω από 19 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν έχουν ένα πρωτεϊνούχο γεύμα κάθε δύο μέρες ούτε κάθε μέρα παραμέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η βοήθεια προς τους πλεοναπόρους. Υπήρχε απόκληση των θέσεων ε, των διαφόρων χώρων μεταξύ τους, αλλά νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια καλή συμβιβαστική λύση, όπου ο καθένας μπορεί να αισθανθεί ότι καλύπτονται οι απόψεις του, με μια κοινή βάση για όλες τις χώρες και με κάποιες σχετικές προσαρμογές. Θέλαμε απλώς να ε, σας ε, επισημάνουμε ένα σημείο που μας, δυσκόλεψε ιδιαίτερος και εκεί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στον κανονισμό, σημειώστε το παρακαλώ, θα το γνωρίζετε, απαγορεύεται, εάν μπορώ να το πω έτσι, απαγορεύεται να λάβει κανείς από φιλανθρωπικές οργανώσεις έστω και συμβολικό ποσό κατά τη διανομή τροφίμων ως βοήθειας που ε, ε, σχετίζονται με τον προέρχονται από το Ταμείο της Βοήθειας προς τους πλειονάπορους. Ε, σας το λέω διότι θα το αντιμετωπίσετε αυτό σε όλες τις περιπτώσεις και τις χώρες. Εδώ δημιουργείται πρόβλημα με τα κέντρα διανομής τα κοινωνικά παντοπολία ε, που τα ποσά αυτά τα λαμβάνουν ως αντάλλαγμα για την διανομή των συγκεκριμένων τροφίμων. Έχουμε ειδοποιήσει την Επιτροπή σχετικά και ο Επίτροπος Άντορ πριν την ψηφοφορία εδώ έκανε μια πολύ σαφή παρέμβαση. Σας το λέω γιατί πραγματικά βρισκόμασταν οριακά στο σημείο που θέλαμε. Η παρέμβαση του Επιτρόπου Άντορ ε, μας επέτρεψε να κρατήσουμε με μεγάλη δυσκολία ανοιχτή αυτή την πόρτα και να συνεχιστεί η λειτουργία των κοινωνικών παντοπολίων. Παρακαλώ λοιπόν να φροντίσετε να διαδοθεί αυτό και να το μάθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Το λέω και υπό τον έλεγχο της Αντριάννα που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, όπου ο Επιτρόπος Άντορ είπε ότι όντως ο κανονισμός ορίζει ότι απαγορεύεται να λάβει κανείς ποσό ω αντάλλαγμα για την διανομή των τροφίμων μέσω του Ταμείου ε, Στήριξης των ε, Πλέον Απορών, αλλά όλες οι άλλες μορφές διανομής τροφίμων που δεν υποφελούνται από το Ταμείο αυτό ακριβώς, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα κοινωνικά λοιπόν ε, παντοπολία βλέπουμε ότι υπάρχουν τρόφιμα να, που μπορεί να προέρχονται από το ταμείο ακριβώς αυτό και άλλα που δεν προέρχονται από εκεί. Μπορούν να συνεχίσουν έτσι να λειτουργούν τα κοινωνικά παντοπολία. Ήταν μια πραγματική δυσκολία αυτή. Και προσπαθήσαμε να την ε, χειριστούμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Δεν ήταν απλό. Πάντω, σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ την Επιτροπή Προπολογισμών. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονε, διότι νομίζω πετύχαμε η πολιτική μας δράση να έχει νόημα και για τους πολίτες και για την Ευρώπη. Ελιζαβέτε, ευχαριστούμε. Ε, ήρθε και στο μεταξύ η Άννη Γένσεν. Αν θέλεις να κάνεις και εσύ κανένα σχόλιο ή να θέσεις και ερωτήματα, διότι έχουμε τις εκπροσώπους εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Πασχόλησης, Γεωργίας και Προϋπολογισμών. Η Έιντερ έκανε μια πρώτη εισαγωγική παρουσίαση. Η Αντριάννα μας έδωσε κάποια στοιχεία, κάποιες απαντήσεις. Θέλεις να παρέμβεις αν ε, σε αυτό το στάδιο συζήτησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει κυρία ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Νομίζω ότι κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη η αλλαγή σε σχέση με αυτό που περιμένουν πολλοί. Εμείς στη Δανία, στη χώρα μου, είχαμε μια πλειοψηφία κατά αυτού του ταμείου. Είπαμε ότι ποτέ ε, δεν πρόκειται να εκταμιευθούν όλα αυτά τα λεφτά. Τελικά μας διέψευσαν οι εξελίξεις και ε, δρομολογούνται προγράμματα με τρόπο ώστε να βοηθηθούν οι πλέον άποροι, αλλά όχι με διανομή τροφίμων. Ε, πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο, αν θέλετε, διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και γι' αυτό σίγουρα το ζήτημα της ε, του να έχουμε μια γενική σφαιρική εικόνα του διαφορετικού χειρισμού από πλευρά των κρατών μελών αυτού του ζητήματος ε, είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Ήταν ε, παλαιότερα ε, τμήμα αυτό τη κοινή γεωργικής πολιτική γιατί είχαμε σοβαρά αποθέματα κρέατο. αυτό δεν ισχύει πλέον. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει και με μια διαφορετική γεύση αν θέλετε και εστιάζουμε πλέον στο τι μπορούμε να κάνουμε για τους απόρους, για να τους ανακουφίσουμε και σίγουρα μόνο που δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε πολλά κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχει γενική άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι κάνουν τα διάφορα κράτη-μέλη, γιατί πιστεύω ότι θα είναι σοβαρές οι διαφορές ε, έχετε στήσει κάποιο σύστημα ανταλλαγή ε, των πρακτικών, ε, διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη χρηστή χρήση των ε, κονδυλίων διότι ξαναλέω ε, η αρχή μου θέση και η θέση της χώρας μου ήταν αρνητική αλλά τώρα τι να πω έχουμε παραδοθεί και βλέπουμε ότι μάλλον είναι καλή ε, η χρήση αυτών των κονδυλίων. Ευχαριστούμε Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ όλους εμπλεκομένους για την πρόοδο που έχουμε επιτύχει και ε, με το Συμβούλιο, διότι τελικά καταλήξαμε στα 3,5 εκατομμύρια ε, για το Ταμείο ε, για το Ταμείο και θα ήθελα τώρα να ρωτήσω κάτι για τα πλεονάσματα, τα γεωργικά πλεονάσματα τι είδους πλεονάσματα έχουμε και τι τα κάνουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και αν υπάρχει καμία δυνατότητα χρήσης ε, αυτών των πλεονασμάτων για τις άπορες οικογένειες. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε τέτοια πλεονάσματα, αλλά να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο. Και ρωτώ, δεν θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να τροποποιήσουμε την νομοθεσία ώστε να το καταστήσουμε αυτό δυνατό. Ξέρω το δικαστήριο μόλις είπε ότι σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία δεν είναι δυνατόν αυτό. Λοιπόν, ρωτώ, με ποιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση να τροποποιήσουμε την ονομοθεσία τόσο ώστε τα παραχθέντα τρόφιμα να χρησιμοποιηθούν. Αυτό είναι κατά της ε, στρατηγικής 2020, της βιώσιμης ανάπτυξης, ε, της ε, αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων, της καταπολέμης, της ένδυας. Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υφιστάμενα γεωργικά αποθέματα και να τα διοχετεύσουμε προς τις οικογένειες που τα χρειάζονται περισσότερο από όλους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Ζωζέ Μανουέλ. Ε, ήρθε και η πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης, ήταν εδώ η Ελιζαμπέτ ήδη, είχαμε αρχίσει να θέτουμε ερωτήσεις ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει της μεθοδολογίας της ομάδας παρακολούθησης γίνεται πρώτα μια ανταλλαγή απόψεων, προκειμένου γιατί για το πρόγραμμα για τους απόρρους της Ένωσης. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι ε, που στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση του προγράμματος και των μελλοντικών προγραμμάτων είναι εδώ για αυτή την ανταλλαγή, τους γνωρίζετε, έτσι είναι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης ε, των τριών γενικών διευθύνσεων απασχόλησης ε, γεωργίας και προϋπολογισμών. Έχουμε, θέλουν και άλλοι το λόγο. Θέλετε, κυρία Μπερές, τώρα το λόγο, όχι στη συνέχεια. Ο Γιάννη Μιλντερ. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια απλή ερώτηση εγώ. Είναι πολύ γνωστό, ευρέως γνωστό, το είπε και η Γιάννη Γιάννησεν ότι δεν είναι ε, από τα 28 κράτη-μέλη όλα κατενθουσιασμένα. Πόσα συμμετέχουν λοιπόν στο πρόγραμμα από τα 28 κράτη-μέλη. Και υποθέτω ότι υπάρχει ένα ποσό που αναλογεί σε κάθε χώρα. Τι γίνεται ε, με το μερίδιο των χωρών που έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια προσέθετα κάτι στην ερώτηση του Γιάν. Από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορείτε να μας δώσετε εσείς μια εκτίμηση, αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο κάθε κράτος μέλος μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα κονδύλια. Δεν λέω να ε, κατονομάσουμε τώρα και να διαπομπεύσουμε καμία χώρα, αλλά να μας πείτε ποιες είναι οι μέθοδοι, αποτελεσματικές, κάποιες λιγότερο αποτελεσματικές ή λιγότερο χρήσιμες. Θα μας ε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Κυρία Τρούπελ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να μάθω ε, το εξή: Όταν κοιτάμε τα διάφορα κράτη-μέλη, Πώς λειτουργεί εκεί η επικοινωνία σε επίπεδο κρατών ακριβώς για να φτάσει στους απόρους αυτή η πληροφορία είναι κοινή η προσέγγιση, είναι διαφορετική ε, στην καθημερινή δουλειά πώς λειτουργούν όλα αυτά. Θα ήθελα λίγη περισσότερη πληροφόρηση σχετικά. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα φυσικά αυτή η ερώτηση. Προσωπικά μπορώ να πω και ε, μιλώ και υπό τον έλεγχο των ε, συναδέλφων μου από τη Γαλλία. Τη μέρα που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε να τερματιστεί το προηγούμενο σύστημα, έγινε αυτό γνωστό στη Γαλλία. Ξαφνικά συνειδητοποίησαν οι Γάλλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθούσε τους απόρους. Άκουσαν, άκουσον. Μέχρι τότε ο Δης ε, είχε επίγνωση αυτού εκτός από την Κατρίνη Τροτμάν. Εντάξει, υπερβάλλω, αλλά όχι πάρα πολύ. Ελάχιστα. Πρόεδρε, αν με επιτρέπετε να σας διακόψω μόνο και μόνο για αυτό το σημείο, και μετά θα περάσω σε γενικότερες τους παρατηρήσεις, αλλά ε, δεν εντοπίζεται τόσο πολύ στον ε, χρόνο, όπως λέτε, η γαλλική θεώρηση των πραγμάτων για την ευρωπαϊκή βοήθεια προς τους απόρους. Έχουμε, είχαμε συνομιλίες ε, με τον Ζακ Ντελόρ και οι Γάλλοι έχουν συγκεκριμένη άποψη για την βοήθεια προς τους απόρους και για την ευρωπαϊκή παρέμβαση σχετικά. Βεβαίως το δικαστήριο έδωσε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση σε όλη αυτή την ε, κίνηση, όμως υπήρχε λόγος που πήρε ευρωπαϊκή διάσταση σε αυτές τις ε, ενέργειες. Ο Κολίος και ο Ντελόρ είναι ακριβώς δύο Γάλλοι που βοήθησαν ακριβώς το να δοθεί μεγαλύτερη προβολή στο θέμα αυτό ε, και στη Γαλλία. Πρόεδρος, ναι, αλλά πριν από 20 χρόνια. Το πρόγραμμα ήταν γνωστό στους Γάλλους, αλλά η συμμετοχή της Ένωσης, που ήταν αρκετά σοβαρή, δεν ε, ήταν τόσο γνωστή. Είναι γαλλογαλλική βέβαια αυτή η συζήτηση και η Χέλγα έχει δίκιο. Θέτει το θέμα του ταμείου και για το ποιε χώρε είναι πιο σοβαρό ή όχι. Κυρία Χόλμαγερ. Έχω κυρίως μια ερώτηση. Σε σχέση με αυτό που είπε ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες. Αν θυμάμαι καλά, και θέλω να ρωτήσω και να μου δοθεί μια απάντηση παρακαλώ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι αν δεν υπάρχουν πραγματικά πλεονάσματα από τη Γεωργία, τότε δεν μπορούν να μεταφερθούν χρήματα από τη Γεωργία για τους απόρους. Αν υπάρχουν πλεονάσματα, τότε βεβαίως τα τρόφιμα που περισσεύουν προφανέστατα μπορούν να δοθούν στον άπορο πληθυσμό. Το θέμα για μας είναι πόσα χρήματα έχουμε τελικά σε αυτό το κορβανά για τους απόρους. Και η δεύτερη ερώτηση. Αυτό το καιρό έχουμε πλεονάσματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε ή πρέπει ή μήπως αυτό το καιρό δεν έχουμε καθόλου πλεονάσματα. Merci, euh, Catherine Ευχαριστούμε κυρία Τροτμάν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ήθελα να θέσω ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα πολύ σύντομη. Υπάρχει, όπως και εσείς το διαπιστώσατε, διαφορά μεταξύ της στιγμής που θα μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στο Ταμείο και της στιγμής που τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τα προγράμματα τους, τα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δράσεις όπου θα συμμετέχουν και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις στη μεταβατική περίοδο. Διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι κατά την περίοδο αυτή δεν θα υπάρχουν και ανάγκες και ότι θα μπορεί να υπάρχει ανάπαυλα στην ε, χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό το σημείο αυτό, ιδίως για την ε, εικόνα που θα δοθεί στους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες φορείς. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, Κατρίν, ο Σαλβατορός Καρίγκα. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω κάτι, μια μικρή διευκρίνηση. Γίνεται λόγο στο Ταμείο αυτό για το δημοσιονομικό κανονισμό που το διέπει. Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποιο τρόπο το Ταμείο αυτό να είναι ad personam και να μην χρειάζεται ειδικό δημοσιονομικό κανονισμό γιατί υπάρχει και ένα διοικητικό κόστος. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Είναι δαπανηρό δηλαδή για να αναπτυχθεί διοικητικά. Το Ταμείο καλύπτει και το διοικητικό κόστος όχι μόνο της αγοράς ε, των τροφίμων από τα πλεονάσματα αλλά και το διοικητικό κόστος της διανομής στα διάφορα Merci Salvador Ευχαριστώ, Γέρον Φέρμ. Ευχαριστώ. στον απόϊχο της παρέμβασης της Αν Γένσεν θα έλεγα και εγώ ότι οι χώρες ε, όπως η Δανία και η Σουηδία ιστορικά ήταν κατά του συστήματος και ο λόγος δεν είναι ότι δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τους απόρους ε, αλλά ότι έχουμε ένα ε, σύστημα πρόνοιας με ένα ισχυρότατο δίχτυ ασφαλείας και δεν συντρέχει λόγος ύπαρξης τέτοιου προγράμματος για τους απόρους. Αυτός είναι ο λόγος. Έχουμε και μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, δεν έχουμε συγγνώμη μη κυβερνητικέ οργανώσει που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα όπω άλλε χώρε ε, και δεν ήταν ξεκάθαρο ο στόχο. Ε, ο στόχο ήταν να βοηθήσουμε του απόλου ή του γεωργού και γι' αυτό στη Σκανδιναβία δεν ήταν δημοφιλέ το πρόγραμμα. Σε σχέση με τον Γιάνν Μόλντερ, ίσω παρανόησα κάτι από αυτά που είπε, αλλά θα μπορούσε να μου το διευκρινίσει. Σε αυτή την κατάσταση με το νέο σύστημα είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν συμμετάσχουν. Δεν υπάρχει ε, περίπτωση opting out ε, μη συμμετοχή ε, σε αυτό το πρόγραμμα. Αν κατάλαβα καλά αυτό που ρώτησε ο Γιάννη Μούλτερ. Ταυτόχρονα υπάρχει όμως και ευελιξία στο ίδιο το σύστημα, από ό,τι κατάλαβα, δεν χρειάζεται ένα κράτος μέλος να χρησιμοποιήσει ε, το σκέλος ε, βοήθειας μέσω τροφίμων. Μπορεί να επικεντρωθεί στα υπόλοιπα σκέλη του προγράμματος ε, και αυτό συμβαδίζει περισσότερο με τα συστήματα πρόνοιας των σκανδιναβικών χωρών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αρμόδιοι να μας, ε, απαντώντας να μας το διευκρινίσουν ε, σε ποιο βαθμό υπάρχει ευελιξία, σε ποιο βαθμό μπορούμε να επικεντρώσουμε τη δράση μας σε κάποια τμήματα του προγράμματος ε, και να επιλέξουμε το opting out για τη βοήθεια με τα τρόφιμα ή κάποια άλλα τμήματα. Υπάρχει περιθώριο ελιγμών για τα κράτη-μέλη. Θα ήταν πολύ σημαντικό να μας το πείτε, διότι από ό,τι ξέρω η Σουηδική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εξετάζει το πώς θα ε, εφαρμόσει το πρόγραμμα και ποια τμήματα ε, θα εφαρμόσει. Ευχαριστώ, Παύλο Ρίμπιχ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για μας είναι πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή να κάνουμε τα σωστά βήματα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ενεργειακή ένδυα. Πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τη θέρμανση και το ρεύμα του. Εκεί τι γίνεται με τα έκτακτα μέτρα και τη βοήθεια προς τους απόρους τους δίνουν φωτοβολταϊκά με μπαταρίες για να έχουν λίγο φως το βράδυ να μπορούν να φορτίζουν τα κινητά τους και τους υπολογιστές. Το έχετε σκεφτεί αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει. Merci bien. Ε, Ευχαριστούμε. Έιντερ, θέλεις το λόγο. Και μετά θα θέσω εγώ ίσως κάποιες ερωτήσεις και υπερβάνεις Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Τροτμάν λίγο με πρόλαβε. Απλώς θέλω να επιμείνω ε, στα μεταβατικά μέτρα λίγο που ρωτούσαμε και στο ερωτηματολόγιο. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά μια συγκεκριμένη ερώτηση. Το 2014 τι θα γίνει τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν πρόκειται να είναι επιχειρησιακά, είναι πλεονασμός βέβαια, λειτουργικά. Δεν θα μπορέσουμε γέρος να δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα. Τι γίνεται από δημοσιονομικής πλευράς, ποια λύση έχετε σκεφτεί, πώς θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό και πώς θα επηρεάσει και τη διαχείριση των ε, ΜΚΟ, των ε, σωματείων των ενώσεων που διαχειρίζονται αυτά τα θέματα, των τραπεζών, τροφίμων, των κοινωνικών παντοπολίων. Τα έχετε σκεφτεί αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είστε και εσείς Πρόεδρος, δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο, αλλά Εδώ λοιπόν νομίζω ότι την ουσία και το περιεχόμενο μπορούμε να τα δούμε μαζί. Διότι αν χρειάστηκε να κάνουμε κάποιους ελιγμούς ε, στην σύνταξη της νομοθετικής ε, πρότασης, χρειάστηκε ακριβώς να συνδυάσουμε τις δύο προσεγγίσεις μας για να συμπληρώσουμε και εμείς τη δική σας. Πριν θέσω κάποιες ερωτήσεις, να τονίσω κάποια σημεία που για μας ως, ε, συντακτών, ως συντάκτες της έκθεσης μαζί σας ήταν της νομοθετικής πρόταση ήταν κάτι πολύ σημαντικό και ήταν σημαντικά σημεία και για μα. Για τα αργιογικά πλεονάσματα λοιπόν. Το κείμενο αυτό παρακολουθεί ακριβώ την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δεν ξανανοίγει το θέμα τη χρήση των γεωργικών πλονασμάτων. Ακριβώ γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα πέρασε από την αρμοδιότητα τη Επιτροπή Γεωργία, ακριβώ στην Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Βέβαια την χάνει η θέση τη Επιτροπή Γεωργία η οποία μας γενοποιηθήκε να λέει ότι τα γεωργικά πλεονάσματα θα έπρεπε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κανείς δεν είναι κατά μια τέτοια προσέγγισης βεβαίως. Συνάδει και με την απόφαση του δικαστηρίου και όχι μόνον. Και με τις προεθέσεις όσων είχαν προσφύγει τελικά στο δικαστήριο. Το ταμείο λοιπόν αυτό δεν είναι ένα ταμείο για την χρήση των γεωργικών αποθεμάτων, αλλά είναι ένα ταμείο κοινωνικής βοήθειας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο για το θέμα της ε, διεύρυνσης του πεδίου ε, του Ταμείου. Σε σχέση με την αρχική αντίληψη για το πνεύμα αυτού του Ταμείου, θέλαμε να υπάρχει διανομή επιστημιστικής βοήθειας και βασικών προϊόντων. Έτσι, το Ταμείο αυτό δημιουργήθηκε ως ε, μία έκφραση της ανησυχίας των κρατών μελών και νομίζω ότι και εσείς το αναφέρατε κυρία Γένσεν έτσι για να ε, καλύψει τις ανησυχίες των κρατών μελών για κάποιους που δεν θέλανε να μιλάμε για την χρήση των γεωργικών προνασμάτων ούτε για επιστηστική βοήθεια. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε μια υποχρεωτική λειτουργία σε κάποιο βαθμό για το ταμείο αυτό ακολουθήσαμε και μια παράλληλη πορεία, δηλαδή την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ή τέλος πάντων την κοινωνική συμπερίληψη, την κοινωνική συμμετοχή και ένταξη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια τελείω διαφορετική προσέγγιση. Όταν καταπολεμά κανεί τον κοινωνικό αποκλεισμό, δεν ελέγχεται, δεν μπορεί να οργανώσει δημόσιες προμήθειες με τους ίδιους όρους που θα το έκανε όπως κάνουν οι τράπεζες επιστημικής βοήθειας που ουσιαστικά μοιράζουν τρόφιμα. Εδώ λοιπόν θέλαμε να έχουμε δύο παράλληλα προγράμματα στο ίδιο κείμενο και το κάθε κράτος μέλος να επιλέξει τη δική του οδό. Αυτή που του αρέσει περισσότερο. Να διαλέξει το δρόμο του για τη δική του τη συμβολή. Τη μια ή την άλλη ή και τις δύο. Πάντως πρόκειται για δύο παράλληλα προγράμματα και ελπίζω ότι αυτό θα καθησυχάσει όσους δεν θέλουν την επισκεπτική βοήθεια, όμως θα πρέπει να ε, συμβάλλουν στο ταμείο αυτό με από άλλη σκοπιά. Τώρα για το θέμα της μετάβασης, της μεταβατικής περίοδου. Βλέπω τις απαντήσεις που μας απέστειλε γραπτός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των διπλωματεύσεων και ότι η αναδρομική επιλεξιμότητα ήταν κάτι που προλάβαμε γιατί δεν έχει ε, καλυφθεί στις βασικές ε, πράξεις της, ε, των διαπραγματεύσεων. Όμως από την, Επιτροπή της, την πλευρά τη Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων χθε μόλις επικυρώσαμε τις σχετικές πράξεις τις κατεξοσοδότηση πράξεις που θα επιτρέψουν ακριβώ την γοργή εφαρμογή τη όλης νομοθεσία. Όμως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει κιόλα τι έχει προβλέψει σε αυτές τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ποιος ακριβώς θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος για τα ποσά τώρα. Το ποσό που, για το οποίο αγωνίστηκε το Ευρωκοινοβούλιο φαίνεται ότι για τον προπολογισμό του 2014 το ποσό θα είναι τελικώς χαμηλότερο χαμηλότερο από αυτό που προέβλεπε η νομική βάση. Ως προς αυτό λοιπόν, εκτός και αν το καλύψατε προηγουμένως, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια περαιτέρω διευκρίνηση γιατί είναι σημαντικό σημείο. Μια διευκρίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι το Κοινοβούλιο επανειλημμένως ψήφισε υπέρ του 3,5, 3,5, αλλά όχι για να το ε, ψαλιδίσουμε στη συνέχεια με λογιστικούς υπολογισμούς. Γι' αυτό λοιπόν θέλαμε να έχουμε μια συγκεκριμένη διευκρίνηση. Αυτά προς τη στιγμή, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε γρήγορα. Γιατί για το Ευρωκοινοβούλιο το θέμα ήταν πραγματικά κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αφορά τους πολίτες. Και γι' αυτό και θέλουμε και την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει σωστή συνέχεια σε όλο το θέμα. Κάτι και ακόμη για τα γεωργικά αποθέματα. Χρειάστηκε να πω ότι δεν είναι πρόγραμμα για, την, για τα γεωργικά αποθέματα, αλλά ενδιαφέρον θα ήταν να το συζητήσουμε και με του υπόλοιπου συναδέλφου. Τι θα γίνει με τα γεωργικά αποθέματα και πώ θα χρησιμοποιηθούν ούτω ή άλλω. Αλλά αυτό είναι μια συμπληρωματική πληροφορία και δεν είναι η βασική μου ερώτηση. Ευχαριστώ, Μπετ. Μετά από αυτές τις ε, Βάσει των πληροφοριών του κ. Δαντάν που είναι στην Επιτροπή Γεωργίας, ε, η χρήση των γεωργικών αποθεμάτων που είναι κάτι ξεχωριστό από το Ταμείο Βοήθειας των Απόρων, Διακόπτει η κυρία Μπερέσα εκτός ε, μικροφώνου. Δεν έχουν σχέση με τα 3,5 ε, δις η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Γκρίλιο Πρόεδρος ε, κανονικά ε, θα μπορεί να μας απαντήσει υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ε, γεωργικά αποθέματα. Α, συγγνώμη, έχουμε και άλλους δύο συναδέλφους που είχαν ζητήσει το λόγο. Η Άλντα πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Ε, μόλις είπε η συνάδελφος Μπερέσε ότι δεν πρόκειται για πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας, είναι ένα πρόγραμμα καταπολέμησης της, του κοινωνικού αποκλεισμού. Το επιβεβαίωσε. Λοιπόν, θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να μας πείτε τι πιστεύετε για τις νέες ανάγκες που υπάρχουν, που δεν είναι επισητιστικού χαρακτήρα, ή μπορεί και να είναι κιόλας, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτό σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν ανάγκες σε διάφορους τομείς για τις πλέον άπορες οικογένειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλλειψη πρόσβασης σε ενεργειακές πηγές, όχι μόνο στο ηλεκτρικό ρεύμα, ε, επίσης ε, πρόσβαση στο πόσιμο νερό ε, και έλλειψη πρόσβαση σε βασικές ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες που έχει οδηγήσει σε χώρες όπως η Ελλάδα ε, σε ε, κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης και κοινωνικής καταστροφής ε, διότι δεν πρόκειται πλέον για μειοψηφικές πληθυσμιακές ομάδες, πρόκειται για σημαντικό τμήμα πολιτών ορισμένων χωρών. Ρωτώ λοιπόν, σε σχέση με τις χώρες που βρίσκονται σε ευπαθέστερη κατάσταση. Θα υπάρξει ε, κάποια ιδιαίτερη διαδικασία στα πλαίσια της υλοποίησης των διατάξεων ε, του προγράμματος του Ταμείου. Ευχαριστούμε. Ρίτσαρτ Άσουορθ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάφορες παρατηρήσεις για τις οποίες ζητώ διευκρίνηση. Ε, κάποιοι συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και εσείς, Πρόεδρε, αναφέρθηκαν στα ίδια σημεία, το λέω εξ Πρώτον, ε, το θέμα των γεωργικών πλεονασμάτων. Ε, τρία πράγματα μου έρχονται κατά νου. Πρώτον, εφόσον μιλάμε για τα αποθέματα, πλεονάσματα μάλλον, δεν ε, υπάρχει καμία αξιοπιστία ή ε, σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλη η διακύμανση ως προς την ποσότητα λόγω της κατάστασης στην παγκόσμια αγορά, στον, στην εποχικότητα της παραγωγής ε, και την η διαθεσιμότητα λοιπόν των πλεονασμάτων δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να υπολογίζουμε. Δεύτερον, η φύση των αποθεμάτων, αν υπάρχουν, πρόκειται, σχετίζεται με βασικά χίδιν αγαθά και δεν πρόκειται για τμήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθεία για επιστημιστική βοήθεια, ε, είτε μιλάμε για δημητριακά είτε για βούτυρο. Δεν μπορούμε να πούμε θα καλύψουμε όλε τι ανάγκε ενό επιστημιστικού προγράμματο. Και τρίτον, ε, ο βασικό λόγο για τον οποίο θα είχαμε ένα απόθεμα παρέμβαση, αν θέλετε να το αποκαλέσετε έτσι, ε, θα ήταν να έχουμε ένα, μια στρατηγική ζώνη απορρόφηση κραδασμών, ούτω ώστε να απορροφούνται τα πλεονάσματα εγκαίρω προτού εκδηλωθεί η έλλειψη. Όμως ε, εφόσον δεν είμαστε στο σενάριο όπως πριν από λίγα χρόνια όπου είχαμε πάρα πολύ ε, μεγάλα αποθέματα, πλεονάσματα βουτύρου, έχει παρέλθει αυτή η περίοδος εδώ και πάρα πολύ καιρό, οπότε ποιο το νόημα. Θα ήθελα λοιπόν να μου διευκρινίσετε στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εντάσσεται πλέον τρόπον την και στην κοινή γεωρική πολιτική. Ρωτώ τους πάντες, ε, η γεωρική πολιτική είναι το σωστό όχημα για να υλοποιούμε κοινωνική πολιτική και αν το κάνουμε αυτό είναι αρκετή η προσθέμενη αξία, δηλαδή σε σχέση με αυτά που δαπανούμε έχουμε ε, ε, το, το προσδοκόμενο όφελος. Ευχαριστούμε. Ρίτσαρτ, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δήλωσε ότι αντιφάσκει με τις συνθήκες η χρηματοδότηση και η προσφορά βοήθεια που έχει γίνει κοινωνική βοήθεια βάσει τη κοινή γεωργική πολιτική. Η λύση αυτή δεν μπορεί πλέον να προκριθεί. Διότι δεν υπάρχουν πλεονάσματα παρά εκτός των εκτάκτων, των εξαιρετικών ε, ετών, με τις εξαιρετικές οδιές, ε, δεν υπάρχει πλεόνασμα γεωργικό. Έτσι λοιπόν με την Επιτροπή και το Συμβούλιο φροντίσαμε να προβλέψουμε και βάσει των ποσών που ως Επιτροπή Προπολογισμών διαπραγματευτήκαμε με το Συμβούλιο για την ερχόμενη επέτεια, Γι' αυτό προβλέψαμε αυτό το πρόγραμμα ως κοινωνικό πρόγραμμα που απευθύνεται στους απόρους. Ο στόχος είναι να τους δώσουμε επισητιστική βοήθεια, αλλά όπως το είπε και η Άλντα, και άλλες μορφές βοήθειας σε τομείς που μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να έχουν σοβαρότατες ανάγκες. Κατά αυτόν τον τρόπο, εάν κάποιες χρονιές υπάρχουν γεωργικά πλεονάσματα, θα δούμε πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά έχουμε αλλάξει άρδιν τη βάση του συστήματος. Ήθελα λοιπόν εγώ ο ίδιος να θέσω κάποια ερώτηση ως συνέχεια ίσως ε, της παρατήρησης που έκανε η πρόεδρος ε, Περβάνος Μπερές για τον προπολογισμό 2014. Τα ποσά δεν συμφωνούν στον προπολογισμό του 2014 ω προς τις πιστώσει πληρωμών, ως τι αναλήψεις υποχρεώσεων με τα 501.300 ευρώ με 1.280.000 για την ε, κοινωνική βοήθεια και όπως γράφεται στο παράρτημα 2 του κανονισμού. Όπως είπε όπως είπε η πρόεδρος Μπερές, το κοινοβούλιο, θέλει η πολιτική αυτή συμφωνία για την επταετία αυτή να τηρηθεί από την πρώτη κιόλας χρονιά, το 2014. Αυτό δεν γίνεται εκτός και αν υπάρξει μια μεταφορά στον προπλογισμό, ένα έμβασμα. μεταφορά πιστώσεων. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι της Γενικής Διεύθυνσης Αποπλαγισμών θα μπορούσαν να μας δώσουν εδώ κάποια διευκρίνηση. Και τώρα να στραφώ στις, ε, στους εκπροσώπους των διαφορετικών υπηρεσιών της Επιτροπής. Ποιος θέλει να κάνει ένα επιπυρός. Αντριάννα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει επέλθει μια πολύ σημαντική αλλαγή στη γενικότερη προσέγγιση. Τι κάνουμε με τους απόρους και τους κοινωνικούς αποκλεισμένους, αυτό το νέο ταμείο. Είναι ευρύτερο το πεδίο εφαρμογή σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας. Επιμένουμε τα κράτη-μέλη όταν δίνουν ε, αγαθά ή τρόφιμα για προσωπική ε, χρήση να παρέχουν και άλλες υπηρεσίες. Δεν θέλουμε απλώς να τους ταΐζουμε εντό εισαγωγικών, αλλά να τους βοηθάμε, ε, να τους παρέχουμε συμβουλές ε, για να μην υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός. Αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή στο νέο σύστημα. Παρακολουθούμε πολύ στενά ε, την ηλική υποστήριξη ε, να συνοδεύεται και ε, υπάρχει και ένα ποσό 5% του συνολικού που να χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη ακριβώ για την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών. Όπως είπε και η κυρία Μπερές, δεν πρόκειται μόνο για διανομή τροφίμων και αγαθών, αλλά και για δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης με ε, πραγματική εστίαση στους αποκλεισμένους, τους απόκληρους της κοινωνίας και τους αποκλεισμένους από την εργασία. Αυτό τι σημαίνει, υπάρχει δυνατότητα, το ανέφεραν ορισμένοι συνάδελφοι, τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν να διανέμουν τρόφιμα να μπορούν να ε, έχουν το δεύτερο είδος ε, επιχειρησιακού προγράμματος και να φτάνουν πραγματικά στους πλέον αποκλεισμένους και να τους βοηθούν να επανεντάσσονται στην κοινωνία και να μην υποφέρουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη τα ίδια να έχουν ε, πλήρη ελευθερία κινήσεων για την απόφαση και ε, ποιες ομάδες στόχους μπορούν να επιλέξουν να περιορίσουν την ομάδα ε, των ενδιαφερομένων, να τη διευρύνουν ή να επιλέξουν κάποιους τομείς ε, και γεωγραφικά που ε, υπάρχει κοινωνική φτώχεια γενικότερα και κοινωνικός αποκλεισμός ή σε όλη την επικράτεια. Αυτό είναι στα χέρια των κρατών μελών. Είναι στη διακριτική τους ευχέρεια. Υπάρχει και εθνική συμμετοχή. Και δεν βλέπουμε κανένα λόγο να μην έχουν όλα τα, κράτη τέτοια προγράμματα συγγνώμη, για να βοηθηθούν οι άποροι στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι όντως ορισμένα κράτη-μέλη δεν επέδειξαν και τεράστιο ενθουσιασμό για τον κανονισμό αυτό, αλλά Δυστυχώς η κατάσταση στην Ευρώπη επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου να βελτιώνεται ο δείκτης της στόχης να μειώνονται τα επίπεδα. Αυτό είναι πάρα πολύ ανισχυτικό και γι' αυτό επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα νέο μέσο, ένα νέο ταμείο που να αφορά όλα τα κρατημέλη και όλους τους απόρους στην Ευρώπη. Ήταν η σωστή απόφαση και ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο που αγωνίστηκε πάρα πολύ σκληρά για να εγκριθεί αυτός ο κανονισμός, έστω και λίγους μήνες μετά την έναξη προγραμματικής περίοδου. Θέλουμε να υπάρξει αλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν διαφορετικά εθνικά συστήματα που μπορούν να υποδεχτούν χρήσιμα αν εφαρμοστούν στα άλλα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει μια πλατφόρμα βάσει του προγράμματος για να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στην ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Ακόμα και μέτρα και δραστηριότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν με μη κυβερνητικέ οργανώσει, εθελοντέ, για να αυξηθεί και η αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Για τα γεωργικά αποθέματα που έγινε μεγάλη συζήτηση, νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε γεωργικά πλεονάσματα. Με την αλλαγή της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής η πιθανότητα είναι όλο και μικρότεροι να υπάρχουν πλεονάσματα που να μπορούν έτσι να διατίθενται και να διανέμονται και γι' αυτό ακριβώς το άρθρο 23 ορίζουμε ότι αν υπάρχουν τέτοια πλεονάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το πρόγραμμα αλλά θα πρέπει να αγοραστούν από το πρόγραμμα. Αυτό ε, προβλέπεται ως ενδεχόν. Ποιος θα τα αγοράσει λέει ο πρόεδρος. Τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν αυτά τα αποθέματα πρέπει να καλύψουν και το λογιστικό κόστος για αυτό. Όχι ο κοινοτικό προπολογισμό. Ε, το ίδιο δεν είναι. Δικό μα προπολογισμό είναι. Είναι 3,5 δις είπαμε. Ε, αν θέλουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματα θα πρέπει και τα πλεονάσματα να τα πληρώσουν όμως. Πολλούνται, δεν διατίθενται. για την ε, επικοινωνία είναι πολύ σημαντικό όντω και τη διαφήμιση. Ε, θα πρέπει και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να τα μαθαίνουν ε, και οι διάποροι. Γι' αυτό στον κανονισμό υπάρχει ειδικό άρθρο που προβλέπει πώς θα γίνεται η επικοινωνία και πώς θα γίνονται γνωστές αυτές οι δράσεις στα κράτη-μέλη. Είναι συγκεκριμένα το άρθρο 19 και είναι από τα πράγματα που θα παρακολουθούμε και εμείς κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων. We uh, Επίσης, έχουμε φροντίσει να καλύψουμε και το διοικητικό κόστος, ένα 5% ενιαίο συντελεστής, γιατί δεν θέλουμε τα κράτη-μέλη και οι ε, οργανώσεις να μπαίνουν στην καθημερινή λογιστική δουλειά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ε, υποστήριξη των απόρων και να μην χαθούμε στις διοικητικές διαδικασίες. Γι' αυτό έχουμε προβλέψει ένα 5% του συνολικού ποσού ε, ως διοικητικές δαπάνες για τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων επιτόπου. Δυνατότητα εξαίρεσης, αυτοεξαίρεσης δεν υπάρχει, out ε, υπάρχει για το γενικότερο πρόγραμμα, για το επισητιστικό υπάρχει. Ξέρω ότι στη Σουηδία έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα και αφορά τους αστέγους. Ήμουν πριν από 15 μέρες εκεί και συναντήθηκα με τους συναδέλφους που εργάζονται πάρα πολύ σκληρά και χαίρομαι που ακόμα και εκείνα τα κρατημέλη που στην αρχή ήταν αναφανδόν κατά της ίδρυσης αυτού του ταμείου τώρα βρήκαν ε, ένα τρόπο να το χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να πιάσουν τον τόπο τα χρήματα. Δεν υπάρχει κίνδυνος να μην απορροφηθούν τα κονδύλια του 2014 γιατί τώρα ισχύουν οι κανόνες των ταμείων συνοχής του νησιν 3. Οπότε οποιαδήποτε ε, δαπάνη του 2014 δεν ε, απορροφηθεί μπορεί να απορροφηθεί εντός της επόμενης τριετίας. Έχουμε τον νησιν 3 παρά τον ετήσιο σχεδιασμό και προγραμματισμό. Έχει μεγάλη σημασία και χαίρομαι ε, που ανισχύει και το Κοινοβούλιο γι' αυτό ότι υπάρχει διαφορά ε, το 11% ε, και των κοντιλιών για το 14. Το είχαμε υπολογίσει με τα 2,5 δισεκατομμύρια. Το ξέρω ότι πρέπει να γίνει μια διορθωτική και συμπροματική πρόταση, αλλά να το προσέξουμε. Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου έχουμε την προθεσμία για να κατατεθούν τα επιχειρησιακά προγράμματα και από εκεί και πέρα έχουμε ένα εξάμεινο για να τα εγκρίνουμε. Δεν θα εξαντλήσουμε το χρόνο μας σίγουρα, ούτε πρόκειται να καθυστερήσουμε κανένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για λόγους ε, προθεσμιών. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και όσο πιο γρήγορα θα προχωρήσουμε. Ξέρουμε ότι είναι επίγουσες οι ανάγκες και επιτακτικές για τα κράτη-μέλη, αλλά... Πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε διορθωτικό και συμπληρωματικό προπολογισμό για να ε, εξασφαλιστούν και για φέτος ακόμα τα κονδύλια. Αν υπάρχει κανένα υπόλοιπο θα το δούμε το 2015. Αλλά το 11% προχρηματοδότησης αρκεί για να καλύψει σχεδόν ένα έτος για την πραγματική εφαρμογή του προγράμματος χωρίς να επιβαρύνει τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Αυτά. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα ε, σημεία. Α, για τις κατεξουδότης πράξεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Απασχόλησης για τη γρήγορη χτεσινή συμφωνία ε, που δεν ε, προέβαλε αντίρρηση και ένσταση με επιστολή. Θα ήθελα να διευκρινίσω υπόψη σας ότι αυτή η κατεξουδότηση πράξη συμπεριλαμβάνει και πρόνοιες για τα συστήματα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου και για τις απαιτήσει αναφοράς. Τώρα είναι στα χέρια των διαχειριστικών αρχών, αλλά για την ε, επιλογή και την επιλεξιμότητα δεν έχει πολύ μεγάλη ε, σχέση. Απλώς είναι τι δεδομένα πρέπει να συλλέγουν και να αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη και με αυτή την κατεξουσιώτηση πράξη δίνουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να προγραμματίσουν σωστά και εγκαίρως. Και η πρώτη έκθεση για αναφορά θα γίνει το 2015. Η αναθεώρηση το 2016, όχι το 2015, για να έχουν ε, αρκετές πληροφορίες στα κράτη-μέλη τι δεδομένα θα πρέπει να συλλέγουν, πώς θα πρέπει να τα διαβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταλάβουμε και πόσο τόπο πιάνει αυτό το Ταμείο τελικά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι μας διαφωτίσατε για πάρα πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό το γεωργικό ε, κομμάτι. Για τα θέματα προϋπολογισμού αναφερθήκατε στο ενδεχόμενο διορθωτικού και συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Μπορείτε, κύριε μου, από πλευράς ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ προϋπολογισμού να μας ενημερώσετε, ναι, Πρόεδρε. με τη στήριξη και την ενεργό δράση του Κοινοβουλίου ε, το πρόγραμμα αυτό αφού απέκτησε νομική βάση μπόρεσε να έχει μια προσάυξηση ε, κατά ένα δις ε, που θα προσθεθεί στα 2,5 δις που είχαν προβληθεί στον αρχικό προϋπολογισμό. Αυτή η αύξηση είναι σε θελούσια βάση των κρατών μελών που κατέθεσαν τα σχετικά προγράμματα. Όπως είπε και συνάδελφος, περιμένουμε τώρα την παρουσίαση των προγραμμάτων κρατών μελών εκ νέου προθεσμία το Σεπτέμβρη και μέχρι τότε ελπίζουμε ότι τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτή τη δαπάνη βάση της νομικής βάσης ε, για το 2014 θα είναι αυτά που επιθυμούμε και ε, ότι ε, θα μπορέσει να γίνει αυτό με μεταφορά Άρα θα χρειαστεί έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ε, δεν θα έχουμε την επαφή διαδικασία του διορθωτικού προϋπολογισμού. Μπορούμε να κάνουμε αυτό το επανομαζομενο fine fine-tuning ε, κατανέμοντας τα επιπρόσθετα ποσά στα σημεία του προϋπολογισμού που τα χρειαζόμαστε. Πρόεδρος, μάλιστα, ε, τα προτιμούμε από όλες τις απόψεις αυτό σαν λύση. Υπάρχει, Πρόεδρε, κάτι άλλο, ερωτήσεις ή από τη δική σας πλευρά, ποιος θέλει το λόγο, ο κύριος ε, Ρικέ. Ε, μία ερωτησούλα που μου έρχεται στο μυαλό. Ε, στην προηγούμενη σύνθεση του προγράμματος, ε, που αν κατάλαβα καλά βασιζόταν στα γεωργικά αποθέματα, αλλά αντιστοιχούσε παρόλα αυτά στα 3,5 δις, ε, υπήρχαν κράτη-μέλη που δεν απορροφούσαν, ενώ τώρα θα απορροφούν όλα, αν κατάλαβα καλά. Ε, η προικοδότηση δηλαδή συνάγω συμπέρασμα για τα μέλη που απορροφούσαν θα ε, μειωθεί. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω με ποιο θαύμα θα εξισορροπηθούν τα ποσά. Δηλαδή, εάν ε, την ίδια πίτα θα τη μοιράσουμε σε περισσότερους, δεν θα έχουν όλοι το ίδιο κομμάτι, άμα καταλάβετε το, το είπα ε, μαθηματικά, λέει ο πρόεδρο είναι προφανή η απάντηση. Πολιτικός πώς τώρα, Περβάνς, μήπω θα μπορούσατε να μα εξηγήσετε για ποιο λόγο ε, επιμείνατε για να είναι υποχρεωτικό το τμήμα. Ναι, απάντηση. Ε, με τη νέα νομική βάση, εξάλλου αυτή είναι η συνέχεια της συζήτησης που κάναμε για τη 2020, για τη στρατηγική 2020 ε, ήταν ολόκληρο ζήτημα. Αν είναι θέμα επικουρικότητας η καταπολέμηση της στόχης ή αν είναι ένα ζήτημα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει. Ε, απόϊχος λοιπόν αυτή τη συζήτηση είναι αυτό που μας απασχολεί σήμερα για το Ταμείο για τους Απόρους, ε, διότι κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι πιο αποτελεσματικό αντίστοιχη δράση να αναλαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο παρότι ε, μέσω ε, παρέμβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρότι ο δημόσιος πολιτικός διάλογος ε, διαρθρώνεται βάσει των ευρωπαϊκών πολιτικών οικογενειών. Λοιπόν, ε, για το Ταμείο για τους Απόρους στον ορισμό είχαμε το ελάχιστο της παρέμβασης ε, των ε, κρατών μελών, ελάχιστος καταμερισμός και αληθεύει ότι τα κράτη-μέλη που βρίσκουμε στο δεύτερο πυλώνα δηλαδή στο πρόγραμμα που σχετίζεται με την κοινωνική ένταξη, είναι ακριβώς οι χώρες που δεν ήθελαν το Ταμείο και άρα πήραν το ελάχιστο ε, απαιτητό στο δεύτερο πυλώνα, ούτως ώστε, με τρόπο ώστε να μην θίγεται το κομμάτι ε, το επισητιστικό. Δεν έχω την κλίδα κατανόμης μαζί μου, όμως πιστεύω ότι στο δημοσιονομικό δελτίο που σίγουρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν αυτές ε, οι πληροφορίες και ξαναλέω αυτές οι χώρες που σας ενδιαφέρουν έχουν τις ίδιες συνθήκες με το προηγούμενο πρόγραμμα, διότι πρόκειται για άλλο σκέλο του προγράμματο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Περβάνω στο Σαλβαντόρ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση και την παρατείνω, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία για την τελική αποτελεσματικότητα. Αν υπάρχουν δύο τρόποι συμμετοχής Ορισμένες χώρες που πιστεύουν στην επικουρικότητα και θέλουν ένα ελάχιστο και κάποιες άλλες χώρες που θέλουν πλήρως να το απορροφήσουν για τη βοήθεια στους απόρους, δημιουργείται εδώ μία αντίφαση μεταξύ, πώς να το πω, της έντασης απορρόφησης ε, ε, του Ταμείου από χώρα σε χώρα και αυτό είναι εις βάρος της τελικής ε, αποτελεσματικότητας. Υπάρχει εδώ μια σημαντική πολιτική συνιστόσα και αυτή η αντίφαση ανάμεσα στην επικουρικότητα και την κοινοτικοποίηση του προγράμματος επηρεάζει άμεσα τη συνολική αποτελεσματικότητα και λειτουργία νομίζω αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί και η Επιτροπή μας εδώ του αλλά και το Κοινοβούλιο συνολικά να ε, ε, ακολουθεί πάρα πολύ στενά ποια θα είναι τα πρώτα αποτελέσματα που θα δώσει αυτό το πρόγραμμα. Ε, μάλιστα, υπερβάσω. Μπορούμε να το ξαναδούμε το θέμα αυτό της νομοθετικής βάσης. Σίγουρα θα υπάρχει τρόπος, δεν ξέρω πώς θα γίνει ακριβώς, αλλά στην, νομική βάση ακριβώς έτσι έχει εγγραφεί. Και ε, αυτό ονομάζεται και το τίμημα μιας πολιτικής, ενός πολιτικού συμβιβασμού. Αλλιώς δεν θα υπήρχε το Ταμείο. Αυτή τη συμφωνία ε, μπορέσαμε να πετύχουμε στο του Συμβουλίου και αποδέχτηκε και το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτήν εγκρίναμε. Όλοι στην Ολομέλεια επικυρώσαμε ακριβώ την ε, νομική βάση για το νέο Ταμείο. Με αυτά τα δεδομένα. Τώρα, ε, ειλικρινώς, εάν Εάν αρχίσω να σκέφτομαι λίγο και να πηγαίνω πίσω στο χρόνο, ε, στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου αποτελείται από ανθρώπου που ήταν υπέρ του Ταμείου, αλλά και από ανθρώπου που δεν ήταν υπέρ του Ταμείου. Συμπεριλαμβανομένου κάποιου που ζήτησε το λόγο και θα πάρει το λόγο να εκφραστεί εντό ολίγου. Όμω αυτή η διαπραγματευτική ομάδα στο σύνολό τη ε, είδε πολύ αρνητικά την συμφωνία ε, στο Συμβούλιο. Διότι ουσιαστικά ε, προβλέπονταν δύο παράλληλα προγράμματα. Όταν καταλάβαμε όμως ότι αυτό είναι το τίμημα για να υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο, το δεχτήκαμε. Το δεχτήκαμε και κοιτάξαμε να επαληθεύσουμε ότι αυτός ο δεύτερος πυλώνας, μου επιτρέπετε πρόεδρε, να αποκαλύψω τελείω το πνεύμα εντό του οποίου εκτελήθηκαν διαπραγματεύσει από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Η δική μα ανησυχία ήταν ότι το τμήμα αυτό, κοινωνική ένταξη, που ζητούσαν οι αντίπαλοι του Ταμείου. Φοβηθήκαμε ότι μπορεί να επικαλύψει ή να ανταγωνιστεί τους σκοπούς ε, λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, διότι στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για πρώτη φορά έχουμε στοχεύσει 20% του προϋπολογισμού που θα πρέπει εφ' να χρησιμοποιείται για δράσεις κοινωνικής ένταξης. Υπήρχε λοιπόν ένα θέμα σύγχυσης των στόχων του ενός και του άλλου ε, μέσου. Ε, γι' αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και γι' αυτό αγωνιστήκαμε, πολεμήσαμε και τα καταφέραμε. Γι' αυτό λοιπόν πετύχαμε να διευκρινιστεί, να διευκρινιστεί στη νομική βάση του ε, Ταμείου για τους πλέον απορούς, ότι το, σκέλος αυτό της κοινωνικής ένταξης θα απευθύνεται ακριβώς στους απόρους και δεν θα συγχαίεται με τις δράσεις που εκτελούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Τώρα, όταν θα δούμε τα δεδομένα που αποβάλλουν τα κράτη-μέλη για να δούμε ακριβώ τι εφαρμόζουν και όταν η επόμενη νέα επιτροπή θα ασχοληθεί καλύτερα ακόμη με τι προποθέσει ε, λειτουργία τη ε, συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τη χρήση του από τα κράτη-μέλη, τότε θα δούμε ακριβώ τι γίνεται από τα κράτη-μέλη βάσει του Ταμείου για του Απόρου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αλλά προβλέφθηκε από τον νομοθέτη ένα πολύ σαφέ όριο μεταξύ των δύο. Ευχαριστούμε, κυρία Κονέλησεν ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ δεν ξέρω αν η κυρία Μπερές εμένα εννοούσε ε, ως αντίπαλο του Ταμείου, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι επί σειρά ετών ήμουν από τους ακριβείς υποστηρικτές του το 2012 όταν στη Γερμανία υπήρξε ε, μάλλον, όταν βγήκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και απείλησε η Γερμανία να σταματήσει το ταμείο, εγώ ε, αγωνιζόμουν για να μην ε, μπλοκάρουν οι κατοχώρες για να σταματήσουν την εμπλοκή ε, στην οποία είχαμε καταλήξει. Γιατί είναι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι άνθρωποι που εξαρτώνται από το προηγούμενο προγράμματο, πρόγραμμα των 25 ετών με τα γεωργικά αποθέματα. Και αυτή είναι για μας η βασική ιδέα ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται βοήθεια. Είναι καλή ιδέα λοιπόν το γεγονός ότι χώρες σαν τη δική μου, οι κατοχώρες ε, ε, συμμετέχει με το ελάχιστο, όπως και η Γερμανία και το Ηνωμένο ε, Βασίλειο, ότι υπάρχουν χώρες με πολύ περισσότερους απόρους που εξαρτώνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το πρόγραμμα. Και αν έπαιρναν το μερίδιό τους όλες οι χώρες, ιδιαίτερα στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες που υπάρχουν οξύτατες ανάγκες και είναι βαθύτατη η κρίση και είναι ε, πολύ ε, άσχημη η ε, φτώχεια και ο κόσμος δεν έχει κυριολεκτικά να φάει, τότε πραγματικά θα λιμοκτονούσαν αν απορροφούσαν οι άλλες χώρες όλα τα δικά τους κονδύλια. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του προγράμματος και υπέρ της εθελουσίας ε, χρήση και στην πράξη εφαρμόζεται σωστά γιατί οι χώρες το έχουν μοιραστεί μεταξύ τους και παίρνουν ε, ανάλογα με τις ανάγκες τους τα κονδύλια που επιθυμούν. Δεν είναι θεωρητικά ή πρακτικά ε, τα προβλήματα και στο προηγούμενο ταμείο ορισμένε χώρε συμμετείχαν, άλλε όχι, ανάλογα με τι ανάγκε του αντλούσαν ε, τη βοήθεια αυτή. Είμαι ε, βέβαιη ότι τα χρήματα ε, πραγματικά θα φτάσουν στους αποδέκτες, τους πραγματικούς απόρους στην Ευρώπη, σε εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Έχουμε δημιουργήσει τώρα ε, επιπλέον δυνατότητες. Μεταξύ αυτών ε, τη διοργάνωση ε, δραστηριοτήτων για να δίνει ο κόσμος τρόφιμα για να μην έχουμε σπατάλες, περιτές, να μην πετάμε τρόφιμα και οι κατασκευαστές και οι διανομείς και οι καταναλωτές να μπορούν να τα δορίζουν στις τράπεζες ε, τροφίμων. Αλλά φοβούμε ότι κάποια κράτη-μέλη που συμμετείχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα απλώς θα συνεχίσουν ε, με την ίδια λειτουργία και θα ε, δαπανίσουν τα χρήματα στις ίδιες ακριβώς δραστηριότητε και δεν θα αξιοποιήσουν ούτε καν θα προσέξουν αυτές τις νέες δυνατότητες. Θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε στην κατάρτιση καλών επιχειρησιακών προγραμμάτων για να τους δώσουμε και μια καθοδήγηση, να μπορούν να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που έχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να πω κάτι σε σχέση με ε, εδώ, αυτά που μας είπε ο Σαλβατόρ. Πραγματικά διαφωνώ. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Οι πολιτικές ε, κοινωνικής ε, πρόνοιας είναι ε, καταρχάς θέμα επικουρικότητας. Είναι διαφορετικά τα συστήματα, διαφορετικά τα επίπεδα και η δομή της φτώχειας. Όλοι έχουν φτωχούς, όμως είναι διαφορετική η κοινωνική διάρθρωση, το μέγεθος και κυρίως είναι διαφορετικά τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό το σύστημα λοιπόν δεν πρέπει να υπερβαίνει ή να αντιβαίνει σε αυτό το εθνικό σύστημα που έχουμε. Χρειαζόμαστε ευελιξία. Είναι απαραίτητη. Εγώ πιστεύω το περιθώριο λίγων θα καταστήσει αποτελεσματικότερο το σύστημα από όταν προσπαθούσαμε να επιβάλλουμε μια ομοιόμορφη λύση για όλους. Θα είναι πιο αποτελεσματικό λοιπόν ε, αν είναι πιο ευέλικτο το σύστημα. Αφήστε που θα γίνει και πιο αποδεκτό σε χώρες που δεν έχουν τέτοια παράδοση. Πραγματικά λοιπόν διαφωνώ με το Σαλβαντόρ και η ευελιξία είναι απολύτως απαραίτητη για να ε, λειτουργήσει ε, εύρυθμα το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε. Ο Σαλβαντόρ. Εγώ δεν έκανα καμιά δήλωση. Απλώς εξέφρασα κάποιους φόβους. Έτσι. Αλλά εντάξει, με κάλυψε ο Γιώραν Φάρμ και διασκεδάστηκαν οι φόβοι μου. Ε, φόβο εξέφρασα, δεν έκανα καμιά δήλωση. So, euh, ο Γιώραν. Άλλες παρατηρήσεις, ε, άλλες ερωτήσεις. Όχι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν απάντησε για την κατανομή του κονδυλίου. Α, ναι, ναι, ναι. Η ερώτηση τη κυρία Κορνέλησεν. Θα απαντήσω στην κυρία Κορνέλησεν, κανένα πρόβλημα. Α, ναι, και του κυρίου Ρικέ την ερώτηση δεν απαντήσατε. Δεν ε, για τα απορρίμματα ε, τροφίμων δεν θα χειριστούμε το ζήτημα μέσα στα επιχειρησιακά προγράμματα. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη να ε, εμπνευστούν από τις πρακτικές όπου τα, για τα απόβλητα τροφίμων, για τις σπατάλη τροφίμων. και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την δυνατότητα για να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με την δυνατή υποστήριξη που υπάρχει για την βοήθεια προς τους απόρους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους δεν ε, περιμένουμε από τα επιχειρησιακά προγράμματα σε καμία περίπτωση να μας πούν πώς τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, χειριστούν το θέμα των πλανασμάτων τροφίμων. Ε, τώρα, ε, υπάρχει ουσιαστική αύξηση. Τα 3,5 δις είναι με τιμές του 11. Δεύτερον, έχουμε 15% εθνική συγχρηματοδότηση για την κατανομή των κονδυλίων του Ταμείου στα κράτη-μέλη. Ε, τα, προ, τα προγράμματα Άγκρη ήταν ε, μέχρι στιγμής ε, χρηματοδοτούμενα 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του προϋπολογισμού που είναι διαθέσιμη για τα επιχειρησιακά θα είναι υψηλότερη για την τωρινή προγραμματική περίοδο. Πρέπει να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι εμπλέκονται όλο και περισσότερα τα κράτη-μέλη και θα συνεισφέρουν στον προπολογισμό και άρα και στη χρηματοδότηση του προγράμματος εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδότηση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την κυρία Μπερέ, την εισηγήτρια, τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΙΔΟΥ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ολοκληρώσαμε την Μέση Διαταξή για την πρωινή συνεδρίαση. Οι συντονιστές να παραμείνουν. και όσοι δεν είναι εδώ παρακαλούν τη βοηθή τους να τους ενημερώσουν ότι προβλέπεται στις 12.30 συνεδρίαση συντονιστών. Θα διακόψουμε ε, για ένα πεντάλεπτο. Ε, μέχρι 12.30 θέλουμε τους διερμηνείς και στις 12.30 θα ε, συνεχίσουμε με την συνεδρίαση των συντονιστών.